διάφορες επιτροπές αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαθεσμικές διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 69 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του ιστορικού κανονισμού. Οι εντολές ε, καταγράφονται στον ιστότοπο της Ολομέλειας. Οι εντολές για τις σχετικέ διαπραγματεύσεις. Και θα ε, δημοσιευτούν και στα πρακτικά τη τρέχουσα συνόδου. Βάσει του άρθρου 69, 4, παράγραφος 2, αριθμός των βουλευτών που μπορούν να ζητήσουν γραπτός μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης 13 Ιουνίου να ψηφιστεί η απόφαση για την άνοιξη των διαπραγματεύσεων πρέπει να συγκεντρωθεί ως τότε και αν δεν υπάρξει τέτοιο αίτημα για ψήφιση στην Ολομέλεια η έναξη των διαπραγματεύσεων θα ε, ξεκινήσει ούτως ή άλλως. Να θυμίσω στην Ολομέλεια ότι την Τετάρτη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψουμε